Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich nehme... Εξαιρετικοί κυρίε και κύριοι, επαναλαμβάνεται η διακοπή σα συνεδρίαση. Ε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η ψηφοφορία για το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης θα γίνει αύριο το μεσημέρι στις 12. Για, ε, πριν περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έχω να σας κάνω δύο ανακοινώσεις. Πρώτον, σύμφωνα με το άρθρο 216 εδάφιο 4 του κανονισμού μας, σας γνωστοποιώ ότι στη διόρθωση που έκανε χτες ε, το απόγευμα η Ολομέλεια στις 5 δεν ζητήθηκε ψηφοφορία οπότε και ε, ούτως εγκρίνεται. Ε, δεύτερη ανακοίνωση. Σύμφωνα με το άρθρο 87α εδάφιο 6